No problem. Good afternoon, everyone. We start. Ξεκινάμε και πάλι με ένα και μοναδικό και μονάκριβο θέμα στην ημερήσια διατάξη που είναι το πρόγραμμα υποστήριξης των δραστηριοτήτων σε ό,τι αφορά την παροχή χρηματοοικονομικών αναφορών και λογιστικού ελέγχου κατά την περίοδο 2014-2020, πρώτη ανταλλαγή απόψεων δίδω το λόγο στον συνάδελφό μου, τον κύριο Στόλογιάν, τον εισηγητή. Ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε. το περιεχόμενο του προγράμματος καταρχήν. Η πρόταση της Κομισιόν έχει προτείνει ένα πρόγραμμα 58 εκατομμυρίων ευρώ για τρεις μη ιδιωτικούς οργανισμούς. Το Διεθνές Ίδρυμα για, την, για τα λογιστικά στοιχεία 32 εκατομμύρια, το Συμβούλιο Παρακολούθηση του Δημοσίου Συμφέροντος 2,3 και η ομάδα ε, χρηματοοικονομικών συμβουλών 23 εκατομμύρια. Ο πρώτος φορέας θα πρέπει να παρακολουθεί από την πλευρά του δημοσίου συμφέροντος τη διαδικασία ανάπτυξης παγκοσμίων ε, προτύπων χρηματοοικονομικών αναφορών και λογιστικού ελέγχου. Οι φορείς αυτοί επίσης συγκεντρώνουν κονδύλια για να χρηματοδοτήσουν το έργο φορέων που θεσπίζουν πρότυπα σε παγκόσμιο επίπεδο. Ο δεύτερος φορέας, η Συμβουλευτική Ομάδα για τις Ευρωπαϊκές Χρηματοπιστωτικές Αναφορές, έχει δύο ρόλους, να δίδει συμβουλές στην Κομισιόν για το κατά πόσο τα λογιστικά πρότυπα, η, η ερμηνεία <clears throat> αυτών των προτύπων συνάδουν με την ε, νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και επίσης δίδει εκ των προτέρων τεχνικές συμβουλές για σχεδιαζόμενα λογιστικά πρότυπα. Είναι μια προορατική δραστηριότητα αυτού του οργανισμού. Γιατί τώρα η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να συγχρηματοδοτήσει αυτούς τους οργανισμούς. Οι παγκόσμιες χρηματοπιστωτικές αγορές χρειάζονται εναρμόνιση των κανόνων λογιστικής και χρηματοπιστωτικών αναφορών σε παγκόσμιο επίπεδο. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για να υπάρξει και μια ολοκληρωμένη αγορά για χρηματοπιστωτικές ε, ε, δραστηριότητες στην Ευρώπη και έχει ζητηθεί να υπάρχει σύγκληση στα θέματα αυτά. Οι χρηματοπιστωτικές αγορές επομένως απαιτούν να υπάρχουν πρότυπα για λογιστική απεικόνηση και χρηματοπιστωτικές αναφορές η Ευρώπη θα χρειαστεί να έχει μεγαλύτερο ειδικό βάρος στη διαδικασία αυτή σε παγκόσμιο επίπεδο, ώστε να είναι ακουστή η φωνή τους. Οι χρηματοπιστωτικές αναφορές και η λογιστική έλεγχη χρειάζονται πρότυπα τα οποία θα πρέπει να αναπτυχθούν επί τη βάση μιας διάφανης και δημοκρατικά υπόλογης διαδικασίας. Και τα διεθνή πρότυπα και οι φορείς οι οποίοι τα θεσπίζουν και οι φορείς οι οποίοι εκπροσωπούν τις ανάγκες της Ευρώπης θα πρέπει να έχουν ανεξαρτησία και επαρκή εμπειρογνωμοσύνη και ικανότητα για να μπορέσουν να παραγάγουν πρότυπα υψηλού επίπεδου και να συμβάλλουν στη διαμόρφωση αυτών των προτύπων και επίσης να έχουν την απαραίτητη οικονομική βάση ώστε να μπορέσουν να εκπληρώσουν το έργο τους προς το κοινό συμφέρον σε μακρόπνο επίπεδο για το 2009-2013 η μεγαλύτερη, η πιο σημαντική δέσμευση ήταν να εφαρμοστεί μια μεταρρύθμιση διακυβέρνησης για αυτούς τους φορείς με στόχο να υπάρξει μεγαλύτερη εμπιστοσύνη των μετόχων, μεγαλύτερη ποιότητα στην ποιότητα των προτύπων καλύτερα και ανάπτυξη αυτών των προτύπων με έναν τρόπο ο οποίος αντικατοπτρίζει το δημόσιο συμφέρον ανεξάρτητα από τη θέληση των επενδεδημένων συμφερόντων. Η Κομισιόν έχει εκδώσει ένα έγγραφο εργασία εκ των προτέρων αξιολόγηση για να υποστηριχθεί η δράση Ευρωπαϊκή Ένωση στον τομέα χρηματοοικονομικών αναφορών και λογιστικών ελέγχων και παρουσιάζει στο έγγραφο αυτό το, τα πορίσματα των μεταρρυθμίσεων διακυβέρνηση. τα θέματα τα οποία πρέπει να τύχουν συζήτηση. Πρώτον, διαδικασία έγκρισης. Η σημαντική σε βάθος χρόνου επενδυτές θέλουν να εξασφαλίσουν από την Κομισιόν την αποτελεσματικότητα της διαδικασίας έγκρισης των προτύπων αυτών για να μπορέσει να εξασφαλιστεί η συμβατότητα μεταξύ του, των προτύπων του IFRS και αυτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Λένε ότι δεν υπάρχει συμβατότητα μεταξύ των δύο ε, ε συστημάτων, των για του Ευρωπαϊκού Νόμου για την ε, ε, λογιστική απεικόνηση και την αντικειμενικότητα που απαιτείται από τα πρότυπα του IFRS σόφρον διαδικασία λογιστικού ελέγχου σημαίνει ότι θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η ανάγκη αποθεματικοποίησης κερδών και διανομής μερισμάτων και επίσης θεωρείται ότι ο μηχανισμός αυτός ο οποίος λειτουργεί μέσω του, της ομάδος εργασίας για τους χρηματοοικονομικούς λογαριασμούς και η δράση των ρυθμιστικών επιτροπών δεν ήταν επιτυχής. Η διαδικασία τώρα είναι η εξής. Οι νέε δομέ στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα εξασφαλίσουν το δημόσιο συμφέρον στο επίπεδο του EFRAG και ESIB. Συζήτησα <laughs> με εκπροσώπους του Διεθνούς Συμβουλίου για την χρηματοοικονομική χρηματοοικονομικές αναφορές, όχι, όχι Συμβουλίου, του Ιδρύματος για τις χρηματοοικονομικές αναφορές και διαφωνούν. Δεν έχουν την διάποψη με αυτά που είπε η ομάδα των επενδυτών. δεν θεωρούν ότι η αντικατάσταση της ε, ε, σοφροσύνης ως έννοιας με την αντικειμενικότητα είναι μια σωστή διαδικασία και συνεχίζονται ακόμα οι προσπάθειες να βρεθεί μια λύση για τα θέματα αυτά. Το θέμα αυτό είναι η υποσυζήτηση λοιπόν ακόμα. Πώς μπορούμε λοιπόν να επηρεάσουμε αυτή τη διαδικασία για τα διεθνή πρότυπα το Συμβούλιο για τα Διεθνή Πρότυπα όλο και περισσότερο έχει διεθνοποιηθεί και εξακολουθεί αυτού του είδους η συζήτηση σε σχέση με την ικανότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να επηρεάσει τη διαδικασία αυτή της θέσπισης προτύπων. με τις βασικές αυτές έννοιες σοφροσύνης ή αντικειμενικότητα. Ένα άλλο θέμα έχει να κάνει με την αποτίμηση των κανονισμών IS. Μάθαμε από τις συζητήσεις με τους εκπροσώπους της Κομισιόν ότι αυτή η αποτίμηση του κανονισμού IAS θα ξεκινήσει σε λίγους μήνες και τα απορίσματά της θα τύχουν αναφοράς τον επόμενο χρόνο. Επομένως, δεν μπορούμε αυτή τη στιγμή να συμπεριλάβουμε και τα απορίσματα αυτά σε σχέση με το πρόγραμμα που έχουμε θέσει σε κίνηση. Υπάρχουν θέματα που άπτονται άμεσα με την πρόταση κανονισμού. Οι χρηματοπιστωτικές πρόνοιες προβλέπονται, όπως σας είπα, 58 εκατομμύρια ευρώ και το ποσό αυτό είναι στο αποθεματικό, είναι υπό επιφύλαξη μέχρι ότου επιβεβαιωθεί ότι είναι συμβατό με το δημοσιονομικό πλαίσιο 2014-2020 αλλά ούτε ο Θεός ξέρει τι μορφή θα έχει αυτό το δημοσιονομικό πλαίσιο μετά τι διαπραγματεύσει από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Εφαρμογή του προγράμματο. Άρθρο 7 τη πρόταση του κανονισμού. Θέλουμε το ετήσιο πρόγραμμα εργασίας, το οποίο εγκρίνεται από την Κομισιόν, να βασιστεί και αυτό στην ανάλυση και αξιολόγηση του προηγούμενου προγράμματος εργασίας. Σε ό,τι αφορά την αξιολόγηση αυτή, η Κομισιόν πρότεινε μία διαδικασία αξιολόγησης και μία έκθεση έξι μήνες πριν από το τέλος του προγράμματος, δηλαδή το 2014 ή νωρίτερα. Για μας θα πρέπει πριν από το τέλος του 2014 να έχουμε μια ε, υποβολή από την Κομισιόν στο Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μια έκθεση για τις απαραίτητες μεταλλαγές στο πρόγραμμα αυτό που προκύπτουν από τη διαδικασία αξιολόγησης του, του κανονισμού IAS, δηλαδή Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα. Προτείνουμε επίσης μέχρι το τέλος του Νοεμβρίου του 2013 και λαμβάνοντας υπόψη τις πληροφορίες που έχουμε πάρει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι ο Επίτροπος Μπαρνιέ θα διορίσει τον Φίλιπ Μάισταντ ως ειδικό σύμβουλο για να προωθήσει υψηλής ποιότητας λογιστικά πρότυπα και δεδομένου ότι αυτός ο ειδικό σύμβουλος έχει σαν καθήκον να παρουσιάσει τελικές συστάσεις για τη βελτίωση αυτής της διαδικασίας προς τον Επίτροπο Μπαρνιέ και τους Υπουργούς στο ΕΚΟΦΗΝ τον Νοέμβριο 2013. Αυτό το οποίο μπορούμε να περιμένουμε είναι να υπάρξει και υποβολή πρόταση έκθεσης από την Κομισιόν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο για τα, για το πρακτέο για να μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε αυτό το πρόγραμμα προς επίτευξη των τεθειμένων στόχων που θα προκύψουν από αυτή την σύσταση. Και επίσης θεωρούμε ότι η Κομισιόν θα πρέπει να υποβάλει και μία έκθεση στη μέση του δρόμου, στη μέση της διάρκειας αυτού του προγράμματος. Αυτά ήθελα να πω και μόνο και με μεγάλη χαρά θα ακούσω τα σχόλιά σας. Και θέλω επίσης να υπογραμμίσω το εξής θέμα. Λαμβάνω χώρα πολλές συζητήσεις και έχω διαβάσει αυτές τις συζητήσεις και έχουμε μια πρόταση κανονισμού που αφορά ένα πρόγραμμα συγχρηματοδότησης αυτών των τριών μη κερδοσκοπικών οργανισμών που ανέφερα προηγουμένω. Φυσικά είναι σημαντικέ αυτέ οι συζητήσει. Από την άλλη πλευρά θα πρέπει να προβούμε σε μια κρίση για το κατά πόσο μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το πρόγραμμα αυτό για να επιτύχουμε αυτό που πιστεύουμε ότι είναι ο στόχος που πρέπει να επιτευχθεί ως αποτέλεσμα αυτών των συζητήσεων διότι κατά τη δική μου κατανόηση δεν είναι και τόσο εύκολο να διαχωρίσουμε τα θέματα αυτά. Δηλαδή τα θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με την συζήτηση σε ακαδημαϊκούς κύκλους, χωρίς να υπάρχει σαφή θέση των εμπλεκομένων και από την άλλη του κανονισμού αυτού, ο οποίος είναι κανονισμός για συγχρηματοδότηση. Σας ευχαριστώ θα μάλα. Ευχαριστώ πολύ λέει ο κύριος Σάλμπα από τους σοσιαλιστές και Δημοκράτης, ο κ. Αλχάντραουι. Ε, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αρχικά να ευχαριστήσω τον εισηγητή για την εκτεταμένη παρουσίαση και φαντάζομαι ότι θα μπορέσουμε να συνεργαστούμε με πολύ καλό τρόπο για αυτή την έκθεση. Πράγματι, μιλάμε για τη στήριξη τριών οργανισμών, τριών φορέων, που και οι τρει διαδραματίζουν πολύ σημαντικό ρόλο στη λειτουργία τη εσωτερική αγορά τη Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και ευρύτερα, παγκοσμίω. Εδώ μιλάμε για ε, επέκταση του υφιστάμενου ε, προγράμματος συγχρηματοδότησης. Είναι λογικό ότι από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από την Επιτροπή ιδίω ε, προσπαθούμε να στηρίξουμε τις εργασίες αυτών των φορέων γιατί θέλουμε να τις επηρεάσουμε. Και έτσι συμβάλλουμε και εμείς σε αυτή τη συζήτηση για να ενισχύσουμε αυτούς τους φορείς. Πέραν της χρηματοδότησης, που είναι απαραίτητη, ε, υπάρχει και ζήτημα δημοσίου συμφέροντος, το οποίο πρέπει να καλυφθεί, γιατί αλλιώς ε, και ιδιωτικοί και άλλοι ενδιαφερόμενοι φορείς θα θεσπίσουν αυτά τα πρότυπα και είμαι πεπισμένος ότι αυτό δεν συμβαίνει πάντα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Έχω όμως ε, ορισμένες παρατηρήσεις. στο Κοινοβούλιο θα πρέπει να ανοίξει μια συζήτηση, να καλέσουμε την Επιτροπή να ε, εστιάσει την προσοχή της σε κάποια σημεία σε ό,τι αφορά τη χρηματοδότηση των φορέων αυτών. Πρέπει να έχουμε μια καλή εικόνα ε, της δράσης τους, ε, του χαρακτήρα τους, των αδυναμιών τους, ελλείψεων, τι μπορούν να κάνουν παραπάνω. Και δεδομένης της κρίσης γίνεται ακόμα πιο σαφής η σημασία της ε, υποβολής εκθέσεων, αλλά και η γλώσσα που διατηρείται ε, σε ό,τι αφορά την χρηματοοικονομική αναφορά. Πρέπει να είναι σαφής λοιπόν οι διατυπώσεις και το ερώτημα που πρέπει να θέσουμε είναι κατά πόσο αυτά τα πρότυπα, οι κανόνες αναφοράς, μήπως είναι ιδιαίτερα περίπλοκοι. Αυτό το e IFRS από ό,τι κατάλαβα χρειάζονται 4.000 σελίδες ε, ε, για να καλυφθεί αυτό το θέμα. Είναι τεράστιος όγκος και η διαφάνεια είναι τμήμα του θέματος. Σίγουρα προβλέπεται αυτό όπως πρέπει, είναι δημόσιες συζητήσεις, αρκεί βέβαια κάποιος να μπορεί να τις καταλάβει. Η ανεξαρτησία τώρα ε, του φορέα απέναντι στον κλάδο, σημαντικό σημείο και αυτό, και ε, σε αυτό το τομέα εργάζεται το IFRS. Πέραν της χρηματοδότησης ε, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό και από τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις που έχουν και τεχνογνωσία, γνώση του πεδίου, αλλά πρέπει να υπάρχουν και εγγυήσει ε, για τη διασφάλιση της ανεξαρτησίας, για να μην υπάρχουν συγκρόμενα συμφέροντα με τέτοιου είδους φορείς. Πρέπει να εξετάσουμε τέτοια ζητήματα σε ό,τι αφορά τα public accounts, τους δημόσιους λογαριασμούς. Ξέρετε ότι υπάρχει ένας εξειδικευμένος φορέας για τον δημόσιο τομέα, όπως και για τον ιδιωτικό. Από το δημόσιο τομέα το θέμα είναι αν θέλουμε να περάσουμε σε έναν ε, φορέα όπως υπάρχει για τον ιδιωτικό τομέα και εκεί υπάρχουν άλλα ζητήματα που εξετάζονται. Θα μείνω εδώ, απλώς ανέφερα κάποια σημεία που θα πρέπει να μας απασχολήσουν, να τα εξετάσουμε. Αλλά δεν νομίζω ότι θα είναι ιδεολογικού περιεχομένου η συζήτηση. Το σημαντικό είναι να λειτουργούν σωστά αυτοί οι φορείς. Ε, ε, επί της αρχής είναι σωστό να τους στηρίζουμε, αλλά θα πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι λειτουργούν και σωστά και ότι υπάρχει διαφάνεια και αποφεύγονται οι συγκρούσεις συμφερόντων. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Αλχαντρόη για τους φιλελεύθερους ο κύριος Κλίντς. Ευχαριστώ πολύ. Μπορώ να επαναλάβω μονάχα αυτά που είπε ο προλαλής σας, ο κύριος Αλχαντραούι, για τη λειτουργία μιας εσωτερικής αγοράς είναι απαράγραπτο να υπάρχουν κοινά πρότυπα για τις χρηματοοικονομικές αναφορές και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει εισαγάγει το 2005 τα διεθνή πρότυπα χρηματοοικονομικών αναφορών ως υποχρέωση των κρατών μελών. Αλλά το ISB, ο φορέας για τα διεθνή πρότυπα στο Λονδίνο, έχει σε μεγάλο βαθμό μια, μια παγκόσμια ακτινοβολία και εμείς είμαστε μειοψηφία εναντί των δικών τους ε, προτύπων. Έχουν αλλάξει λιγάκι τα πράγματα, έχει μειωθεί κάπως η επιρροή των Αμερικανινών από ό,τι καταλαβαίνω και κάπως έχει αυξηθεί η επιρροή των Ευρωπαίων. Αλλά ακόμα δεν υπάρχει αυτή η ισορροπία η οποία έπρεπε να υπάρχει και θα πρέπει να κατανοήσουμε ότι όπως και στο παρελθόν οι Ηνωμένε Πολιτείε δεν είναι έτοιμες να ε, αλλάξουν πορεία και να υιοθετήσουν το IFRS. Η δική μας ελπίδα, εγώ το 2004 στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τότε ο, ο πρεσβευτής των ΗΠΑ, ο Αλεξάνδρου Σάου, μου είχε πει αυτό είναι θέμα ε, μηνών, αλλά μετά από 10 χρόνια σχεδόν εξακολουθεί να είναι ευσεβής πόθος και μόνο αυτή η πρόθεση να, αποδεχθεί, να αποδεχθούν οι ΗΠΑ Πολιτείες το IFRS. Επομένως, αυτό το οποίο είναι απαραίτητο είναι και εμείς να εξασφαλίσουμε ότι και εμείς έχουμε μια καλύτερη κατανόηση για το ISB. Εγώ φυσικά θέλω να έχουμε το IFRS ως ε, παγκόσμιο πρότυπο και όχι να το αντιμετωπίζουμε μονάχα σαν αποκλειστικά ευρωπαϊκό, γιατί αυτό θα έχει αντιπαραγωγικό χαρακτήρα. Θα πρέπει να ξέρουμε ότι χώρες όπως η Κίνα, η, Κίνα, η Ιαπωνία, το Μεξικό και άλλες χώρες Βασιλεία που είναι έτοιμες να μπουν σε αυτά τα πρότυπα <clears throat> και αυτές θα πρέπει να συμβάλλουν στη διαδικασία εξέλιξης αυτού του <clears throat> προτύπου. Επομένως θα πρέπει και εμείς να παίξουμε και ένα χρηματοδοτικό ρόλο για την εξέλιξη αυτών των προτύπων. Δεν είμαστε μόνοι μας λοιπόν και θα πρέπει να μας ε, ενδιαφέρει ο συνολικός προϋπολογισμός που δίνουμε εμείς ως μερίδιο στο συνολικό προϋπολογισμό αυτών των Ιδρυμάτων. Και ποιο είναι το ειδικό μας βάρος ως ποσοστό στη, σε σχέση με τους άλλους ε, χρηματοδότες. Έχουμε λοιπόν το απαραίτητο οικονομικό ειδικό βάρος μέσα σε αυτούς τους οργανισμούς οι οποίοι παράγουν τα πρότυπα. Δεύτερον, καταλαβαίνω ότι υπήρξε μια ιστορική πορεία, αλλά είναι τεράστιος ο αριθμός των φορέων που ασχολούνται με το ίδιο αυτό θέμα. Όταν βλέπω πώς οι μεμονωμένοι φόροι, συμβούλια, καταπιστεύματα ασχολούνται με αυτά τα θέματα, αρχίζω να ζαλίζομαι. Και αναρωτιέμαι μήπως θα μπορούσαμε να ξεκινήσουμε από το μηδέν πάλι, να δούμε με ποιο τρόπο θέλουμε να οργανώσουμε τα πράγματα, να ξεκινήσουμε δηλαδή από μια νέα εκκίνηση και ενδεχομένως να τα βγάλουμε πέρα με το ένα δεύτερο μονάχα των φορέων που δραστηριοποιούνται στο, στο θέμα αυτό. Όλα αυτά δεν βοηθούν λοιπόν την πραγματικότητα και την πρόοδο των προτύπων. Εν πάση περιπτώσει έτσι ιστορικά έχουν εξελιχθεί τα πράγματα και δεν είναι εύκολο από τη μια μέρα στην άλλη να τα αλλάξουμε όλα αυτά. Αυτό το οποίο για μένα είναι αποφασιστικό είναι το θέμα του μελλοντικού ρόλου της ΕΦΑΚ και της PIOB, δηλαδή τον, ε, το ρόλος του Ιδρύματος ISB είναι σαφής. Αλλά το θέμα γίνεται, το θέμα τώρα είναι πώς, ποιος θα αποτελέσει το φορέα παροχής συμβουλών για την Κομισιόν, για το οποίο η το ερώτημα είναι με ποιο τρόπο θα πρέπει να προχωρήσουμε στο μέλλον, θα πρέπει να κατανοήσουμε ότι για την ε, οδηγία που αφορά τους ε, ορκωτούς λογιστές θα κληθούμε να αποφασίσουμε τον Ιούλιο και επομένω θα πρέπει να δούμε πώς γίνεται η όλη διαδικασία της εποπτείας των ορκωτών λογιστών στο μέλλον. Και πρέπει να θέσουμε και το ερώτημα με ποιο τρόπο θα πρέπει να εξασφαλίσουμε τη χρηματοδότηση της PIOB μέχρι να φτάσουμε σε τελικό επίπεδο σε αυτή τη διαδικασία. Και εδώ η εποπτική αρχή για τις ε, ε, χρηματαγορές και χρηματιστήρια θα πρέπει να παίξει κάποιο ρόλο κατά την απόψη μου. Ε, αυτό το οποίο είναι σαφές είναι ότι θέλουμε να έχουμε κοινά πρότυπα για τους λογιστικούς ελέγχους και τις ε, χρηματοοικονομικές αναφορές, αλλά de facto δεν έχουμε τέτοια κοινά πρότυπα. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Για τα κρατικά ομόλογα όταν έχουμε μια χώρα περιφερική, παραγωγή η οποία βρίσκεται σε δυσκολία και η οποία ε, πουλάει τα ομόλογό τη σε τρεις χώρες και σε τρεις διαφορετικές τράπεζες. Είναι διαφορετική αντιμετώπιση. Αλλού θεωρείται ότι είναι το 22% της ονοματικής αξίας που θα πρέπει να τιμή αγοράς, άλλοι λένε 55%. Επομένως, έχουμε την, ε, το ίδιο αξιόγραφο το οποίο αντιμετωπίζεται τόσο διαφορετικά από διαφορετικούς λογιστικούς ελεγκτές. Μια χώρα λέει ας πούμε ότι αυτό είναι το 22% της πραγματικής αξίας, η άλλη 55%. Εδώ έχουμε μια τεράστια διαφορά. Είναι δυόμιση φορές διαφορά από τη μία κρίση στην άλλη. Εδώ έχουμε λοιπόν πολλή δουλειά μπροστά μας. Αυτό το οποίο είναι σημαντικό να εξασφαλίσουμε ότι και οι οργανώσεις ομπρέλας που έχουν να κάνουν με τους ε, ε, οικονομικούς ελεγκτές θα πρέπει να έχουν κάποια κοινά πρότυπα και αυτό έχει μεγάλη σημασία για μας. Ένα τελευταίο σημείο και έχει αναφερθεί σε αυτό ήδη ο εισηγητής μας. Ο κανονισμός IAS και η αναθεώρησή του είναι κάτι που έχει υποσχεθεί ο Επίτροπος Μπαρνία εδώ και ένα χρόνο, το Μάρτιο του 2012, αυτό το οποίο πρέπει να εξασφαλίσουμε. Είναι ότι κάποτε θα λάβει χώρα και θα, αυτή η μεταρρύθμιση. Τώρα που έχουμε τη συνδίκη της Λισαβόνας και νέους κανόνες, δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί σαν να μην υπάρχει η συνδίκη της Λισαβόνας, θα πρέπει να υπάρχει προσαρμογή στις νέες θεσμικές συνθήκες. Ευχαριστώ κύριε Κλίντς για τους πράσινους. Ο κύριος Γκίνγκολτ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Θα ήθελα να προβώ σε κάποιες παρατηρήσεις. Ευχαριστώ για αυτά που είπατε. Τα περισσότερα θέματα εκαλύφθησαν ήδη από τον εισηγητή, αλλά και από συναδέλφους. Αυτή η έκθεση είναι τόσο ενδιαφέρουσα διότι μας δίνει τη δυνατότητα να συζητήσουμε ξανά, όπως είπε ο Βόλφ, διότι δεν είναι κοινή συζήτηση, να συζητήσουμε ξανά πώς σχετίζεται η Ευρώπη, η Ευρωπαϊκή Ένωση με παγκόσμιους φορείς που καθορίζουν τα παγκόσμια πρότυπα. Μας συμφέρει να έχουμε παγκόσμια πρότυπα. Και χρειαζόμαστε συγκρίσιμα πρότυπα σε πολλούς τομείς. Γι' αυτό συμφωνώ με το Βόλφ και με τους άλλους που είπαν ότι εδώ εμπεριέχεται μία αξία, αυτή καθ' αυτή. Ακόμα και αν υπάρχει ιστορική εξέλιξη στις δομές και δεν υπάρχει κάποια συγκεκριμένη προσέγγιση προς δημιουργία παγκοσμίων φορέων και παγκοσμίων προτύπων, παρόλα αυτά πρέπει να τα δημιουργήσουμε. Το βλέπουμε σε διάφορα σχήματα. Κάποια σχήματα βασίζονται στον ΟΗΕ, άλλοι μηχανισμοί στην Επιτροπή της Βασιλείας, που είναι άλλη δομή. Η ΑΙΟΣΚΟ έχει ένα άλλο ιστορικό. Με το ISB έχουμε άλλο σύστημα. Και με τους άλλους οργανισμούς υπάρχει διαφορετικό ιστορικό, αυτούς που αναφέρθηκαν. Αυτό δεν θα μπορέσουμε να το αλλάξουμε εν μία νυχτή. Και δεν θα μπορέσουμε να εφαρμόσουμε συγκεκριμένους κανόνες που θα είναι μέτρο δικό μας, μέτρο στάθμισης δικό μας στην Ευρώπη, να το εφαρμόσουμε σε παγκόσμιο επίπεδο. Εμείς θέλουμε δικές μας αρχές, δημοκρατία, λογοδοσία, διαφάνεια και ούτω καθεξής. Αυτές είναι οι βασικές ιδέες ε, του κράτους δικαίου. Αυτό δεν υπάρχει στο παγκόσμιο επίπεδο, διότι δεν έχουμε παγκόσμιο κράτος. We will not be able Γι' αυτό δεν θα μπορέσουμε να εφεύρουμε από την αρχή ένα παγκόσμιο κράτος. Προφανώς βέβαια θεωρητικός στόχος θα πρέπει να είναι να κινηθούμε σε αυτή την κατεύθυνση. Ούτως ώστε συμβάλλουν και οι Ευρωπαίοι να δημιουργηθούν θεσμοί που να ταιριάζουν με αυτά τα πρότυπα. Που σε μεγάλο βαθμό θα ενστερνίζονται τα θεμελιώδη δικαιώματα που γίνονται αντιληπτά σε παγκόσμιο επίπεδο. Θα επικεντρώσω την παρέμβασή μου στο ISB. Το ISB παράγει δημόσια αγαθά παγκοσμίου εμβελίας. Δεν είναι κάτι ιδιωτικό, διότι τα λογιστικά πρότυπα ε, είναι παγκόσμια δημόσια αγαθά ως κανόνες επισκεφτήκαμε το ISB, ήταν ενδιαφέρουσα επίσκεψη, πήγαμε το Δεκέμβριο με τον συνάδελφο Όλε Σμιτ και με τη γραμματεία. Πολύ ενδιαφέρουσα επίσκεψη. Μας υποδέχτηκαν πολύ ε, αξιοπρεπώς, μας ετίμησαν, αλλά ήταν μια εμπειρία που δεν θα λησμονήσω. Συναντηθήκαμε με το Παγκόσμιο Διοικητικό Συμβούλιο του ISB, Έγινε πολύ ενδιαφέρουσα ανταλλαγή απόψεων. Απ' την άλλη, είδα ότι υπήρχε μεγάλη αυτοπεποίθηση για αυτό τον οργανισμό σε σχέση με, δημοκρατικό, με το δημοκρατικό τρόπο λειτουργίας. Και η νοτροπία με ενδιαφέρεται. Τα μέλη εκπροσωπούσαν κατά κάποιο τρόπο τις χώρες τους, βέβαια, όχι τα κράτη αυτά κάθε αυτά, εκπροσωπούσαν μια γεωγραφική περιοχή μια... και πώς είχαν επιλεχθεί. Και υπήρχε μια γεωγραφική ισορροπία. Λοιπόν, εμείς σαν Ευρωπαίοι θα πρέπει να διερωτηθούμε. Σε ποιον λογοδοτούν αυτοί που εκπροσωπούν τις ευρωπαϊκές περιοχές. Δεν θα περίμενα οι Κινέζοι, ο Κινέζος εκπρόσωπος να εκλέγεται δημοκρατικά. Παρ' όλα αυτά θέλουμε να συνεργόμαστε στο παγκόσμιο προσκήνιο. Δεν μπορούμε να πετήσουμε δημοκρατία για όλους, προφανώς οι Ευρωπαίοι εκπρόσωποι. Όμως, ο εκπρόσωπος που είναι στο Συμβούλιο εκεί, γιατί προέρχεται από την Deutsche Bank, αυτός που εκπροσωπεί τη Γερμανία, με εξέπληξε. Όχι ότι έχω κάποιο πρόβλημα διότι κάποιος που προέρχεται από την Deutsche Bank δεν είναι ο ενδεδειγμένος, αλλά στην Ευρωπαϊκή μια ευρωπαϊκή χώρα θα πρέπει να εκπροσωπείται από κάποιον μετά από μια ανοιχτή διαδικασία επιλογής και κατόπιν δημοκρατικής αποφάσεως. Αυτό το βρήκα πολύ ενδιαφέρον. Και κάτι άλλο ήταν ενδιαφέρον. Πώς διεξάγονται οι συζητήσεις. Το πρότυπο της διαφάνειας, τι να πω, ε, τα πρότυπα που χρησιμοποίησαν τη διαφάνεια ήταν πολύ λογικά. Αν προτείνεται ένα πρότυπο, ανεβαίνει στην ιστοσελίδα, μπορεί να σχολιάσει οποιοδήποτε, δημόσια προσέγγιση, διαφάνεια, ποιο σχολιάζει, τι λέει, και μετά λαμβάνεται μια απόφαση των αρμοδίων φορέων. Και κάτι άλλο που βρήκα ενδιαφέρον. Όσον αφορά τη διαφάνεια, όλοι είναι ίσοι. Αν κάποιος λογιστής κάπου, ας πούμε στις νήσους Κουκ, έχει κάποια άποψη, η γνώμη του έχει την ίδια, το ίδιο βάρος σαν να είχε πάρει απόφαση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ακόμα και αν ένα διεθνές κοινοβούλιο, σαν το δικό μας, ζητήσει κατά χώρα Φερρυπίν αποβολή αναφορών και δεν μοίραμε απάντηση ούτε μετά από τρία χρόνια ο κ. Χούγκεφορς, ο πρώην πρόεδρος, ε, δεν απάντησε. Όταν μπήκε ο καινούριος πρόεδρος μας, απάντησε μετά από τρία χρόνια. Ερώτηση. Ποιος αντιμετωπίζεται πώς. Η διαφάνεια όσον αφορά τον προπολογισμό άλλο θέμα. Η Ευρώπη πληρώνει πολλά, πληρώνουμε πολλά και μας ζητείτε να πληρώσουμε ξανά πολλά χρήματα. Και ένα ερώτημα που τίθεται είναι αυτό που έθεσε ο Βολφ Κλίμτς. Πόσα πληρώνουν οι άλλοι. Υπάρχει αναλογικότητα. Δεύτερο ερώτημα. Τα χρήματα καταβάλλονται ανάλογα με την επιρροή που έχουμε. Τρίτον, ποιος άλλος πληρώνει. Από ό,τι έμαθα στην επίσκεψη, φαίνεται ότι οι μεγάλες τέσσερις λογιστικές εταιρείες πληρώνουν πολλά, μεγάλο ποσοστό του προπολογισμού. Δεν ξέρω ποιος πληρώνει πόσο, θα ήθελα να ξέρω λεπτομέρειες και θα ήθελα να ξέρω πόση επιρροή πετυχαίνουν αυτοί με τα ποσά που πληρώνουν. Τέλος. Πρέπει να δούμε θετικά αυτούς τους οργανισμούς καταρχήν. Θέλουμε παγκόσμιας εμβέλειας φορείς, αλλά σαν Ευρωπαίοι πρέπει να θέσουμε τα ερωτήματά μας βάσει των αξιών μας. Δηλαδή δημοκρατικός έλεγχος, διαφάνεια. Αν χρησιμοποιήσουμε δημόσια χρήματα που καταβάλουν οι πολίτες βάσει δημοκρατικών αποφάσεων, τι παίρνουμε για αυτά τα χρήματα που πληρώνουμε. Δεν αρκεί κατά την άποψή μου να υπάρχει ένα συμβουλευτικό φορέα που μπορεί να πηγαίνει από καιρού καιρών ο κύριο Μπαρνιέ. Τον σέβομαι τον κύριο Μπαρνιέ, δεν λέω. Αλλά κανονικά με τα χρήματα πρέπει κάποιο να... να πετυχαίνει το ότι οι εκπρόσωποι τη Ευρώπη θα εκπροσωπούν τι αξίε μα, θα επιλέγονται βάσει δημοκρατικών αξιών. Καλή στιγμή λοιπόν τώρα ε, να συζητήσουμε με αυτού του φορεί πρότυπα Πώς θέλουμε οι ευρωπαϊκές αξίες και οι ευρωπαϊκές αρχές για την παραγωγή δημοσίων αγαθών να χρησιμοποιούνται. Πολλοί υπέφεραν στην Ευρώπη για τη δημοκρατία αυτές τις αξίες. Ο κόσμος πολέμησε για αυτές τις αξίες. Και όταν κινηθούμε στο παγκόσμιο επίπεδο, θέλουμε κάτι να αντιστοιχεί σε αυτά που καταβάλουμε και να υπάρχει μια αντιστοιχία στο προϊόν που παράγεται που σχετίζει τις βασικές αξίες μας. Θα πρέπει να γίνουν αυτές συζητήσει με και ίσως με συμμετοχή αυτών των φορέων. Να συζητήσουμε και οργανωτικές αλλαγές που θα αντιστοιχούσαν σε αυτές τις αξίες που προανέφερα. Σταματώ εδώ. Προσβλέπω σε μία άκρο ενδιαφέρουσα έκθεση. Κύριε Στόλογιαν, σας θαυμάζω για αυτό που κάνατε. Πραγματικά ενδιαφέρον ο ρόλος να δημιουργεί κανείς κάτι τόσο που είναι θεσμούς οι οποίοι είναι πιο ελέγξιμοι και που αντιπροσωπεύουν παγκόσμιες τέτοιες αξίες. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Γκίγκολτ για τους συντηρητικού και μεταρρυθμιστές. Ο κύριος Στέγιακ. Πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση και ο, η συζήτηση, η ομιλία του συναδέλφου εγώ εκπροσωπώ τον ε, Σκιώδη από πλευράς ε, ECR. Επομένω θα προσπαθήσω να διαβάσω στα αγγλικά. Τον τελευταίο χρόνο, λέει λοιπόν ο κύριος Καμάλ, ήρθα σε επαφή με αριθμό επενδυτών που έχουν εκφράσει επιφυλάξεις και ανησυχίες για το συνεχιζόμενο πρόγραμμα για τη δημιουργία διεθνών ε, προτύπων χρηματοοικονομικών αναφορών. Εγώ συμμερίζομαι τις ανησυχίες τους ότι οι ευρωπαϊκοί και αμερικανικοί ε, ε, λογαριασμοί εξυπηρετούν σχετικά διαφορετικούς στόχους και υπάρχει κίνδυνος να υπάρξει σύγχυση μεταξύ των δύο συστημάτων. Στις ΕΠΑ οι λογαριασμοί από το 1993 που εισήχθη αυτό το σύστημα ε, εξυπηρετούν ε, έναν στενότερο στόχο, δηλαδή την παροχή πληροφοριών ε, για τις υπηρεσίες τέτοιων επιχειρήσεων στην αγορά. Στην Ευρώπη πάμε πολύ πιο πίσω και τέτοιου είδους υπηρεσίες συνδράμουν σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό στην διακυβέρνηση, στην οικονομική διακυβέρνηση. Τέτοιοι λογαριασμοί μπορούν να υπογραφούν μόνο από ελεγκτές για να διασφαλιστεί ότι ε, προστατεύονται τα συμφέροντα των, ε, ε, των επενδυτών. Τα τελευταία 30 χρόνια το Διεθνές Πρόγραμμα Σύγκλησης, το οποίο συντονίζει ο IASB, δείχνει ότι υπάρχει, υπάρχει συμβιβασμός, αποδυνάμωση και φαίνεται ότι τα διεθνή πρότυπα που έχουν δημιουργηθεί και εισαχθεί από το 2002 στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ε, ίσως ε, υιοθετήθηκαν ε, εσφαλμένα. Τα IFRS μπορούν να υιοθετηθούν μόνο αν πληρούν τα κριτήρια του Ευρωπαϊκού Εταιρικού Δικαίου. Πρέπει λοιπόν να συζητήσουμε επί του ρόλου που θέλουμε να διαδραματίσουμε, διαδραματίσουν τέτοιοι λογαριασμοί στην Ευρώπη. Ε, η εκτίμηση στοιχείων του ενεργητικού υπαθετικού ε, ανά κάποια χρονική στιγμή, τότε εντάξει. Αν όμως θεωρούμε ότι πρέπει οι λογαριασμοί αυτοί να δίνουν κίνητρα στους ε, διοικητές και διευθυντές ε, να λειτουργούν τις επιχειρήσεις τους προς όφελος των καταναλωτών και επενδυτών, τότε η προσπάθεια προσύγκληση πρέπει να συνεχιστεί. Εγώ είμαι υπέρ της διεθνούς ε, σύγκλησης ε, ε, σε ό,τι αφορά τα πρότυπα, όμως δεν μπορώ να στηρίξω αυτό το project, αυτό το πρόγραμμα, εάν το αποτέλεσμα είναι σύγκληση προς κακής ποιότητας πρότυπα, που δεν πληρεί τις προϋποθέσεις του ευρωπαϊκού δικαίου. Αυτά λέει ο κ. Καμάν. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Δεν ξέρω αν η Επιτροπή θα θέλει να λάβει το λόγο. Παρακαλώ. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Ακούσαμε μία σειρά από παρεμβάσεις και τις ανησυχίες, τις βασικές ανησυχίες των μελών της Επιτροπής σας για τα κύρια ερωτήματα τα οποία πρέπει να αντιμετωπιστούν τους επερχόμενους μήνες. Ε, Έχουμε ακούσει για τη διαδικασία αξιολόγησης που έχει προτείνει ο Επίτροπος Μπαρνιέ και η οποία αυτή τη στιγμή γίνεται στη Γενική Διεύθυνση Αγοράς. Υπήρξε μια <clears throat> διαδικασία υποβολής προσφορών για την εκπόνηση αυτής της μελέτης και ελπίζουμε ότι στα μέσα του 2014 θα έχει τελειώσει αυτή η διαδικασία. Έχει ξεκινήσει επομένω. Επίσης αναφερθήκατε στην αποστολή η οποία έχει δοθεί στον κύριο Μέιστάτ από τον Επίτροπο Μπαρνιέ ο στόχος μετά από τις συζητήσει που έγινε στο Συμβούλιο Κοφίν του Νοεμβρίου 2012 ο στόχος είναι να μπορέσει να τεθεί το ερώτημα του πώς <clears throat> μπορούμε να συμβάλλουμε αποτελεσματικά στις διαδικασίες αυτές τυποποίησης σε παγκόσμιο επίπεδο. Έχουμε πολλούς ε, φορείς, το ΦΡΑΚ, το Συμβούλιο του Τεχνικό της Κομισιόν, το ΑΡΚ, την Επιτροπή των Κρατών Μελών για τα θέματα αυτά. Πώ λοιπόν θα μπορέσουμε να συντονίσουμε όλου αυτού του φορεί για να μπορέσουν να γίνουν ακουστέ οι απόψει μα στο ISB. Η αποστολή αυτή αναλαμβάνεται από τον κύριο Μέιστατ τώρα και στο τέλος Νοεμβρίου περιμένουμε τα πορίσματά του. Περιμένουμε λοιπόν από τον κύριο Μέιστατ σημαντικές απαντήσεις σε αυτά τα ερωτήματα. Μιλήσαμε για την έννοια της επιφυλακτικότητος ή της προληπτικότητος έναντι της ε, ουδετερότητος. Είναι αυτές έννοιες οι οποίες αναφέρονται σε σχέση με το ενιολογικό πλαίσιο του ISB. Είναι ένα σημαντικό πλαίσιο, το οποίο όμως και αυτό είναι υπό αναθεώρηση. Το ISB έχει ξεκινήσει μια διαδικασία αναθεώρηση αυτού του ενοιολογικού πλαισίου και αυτή είναι η στιγμή για την οποία, κατά την οποία θα πρέπει να επανέλθουμε και να εξετάσουμε όλε αυτέ τι έννοιε. Αυτό είναι το χρονοδιάγραμμα λοιπόν. Έχουμε όλα αυτά τα ενεξέλιξη σχέδια. Θα ήταν ε, σωστό λοιπόν να περιμένουμε να έχουμε τις απαντήσεις και να ακολουθήσουμε τη σωστή χρονική σειρά. Τώρα βέβαια το τωρινό χρηματο δημοσιονομικό πλαίσιο εκπνέει στο τέλος του 2013 και αν θέλουμε να διατηρήσουμε την ευρωπαϊκή επιρροή στους φορείς αυτούς, ιδίως αν θέλουμε να αυξήσουμε περισσότερο, η Κομισιόν θεωρεί ότι θα πρέπει να διατηρήσουμε αυτή τη χρηματοδότηση, ιδίως σε επίπεδο του ISB, ώστε το εποπτικό του Συμβούλιο για να εξακολουθήσει να είναι μέλος του Επίτροπος Μπανία πρέπει να συμβάλλει και η Ευρωπαϊκή Ένωση στην χρηματοδότηση του ISB. Τα άτομα λοιπόν τα οποία θεσπίζουν, τα οποία συγγράφουν και θεσπίζουν τα πρότυπα πρέπει να έχουν μια ισορροπία σε σχέση με την προέλευσή του, σε σχέση με τη γεωγραφική του προέλευση, να μην είναι μονάχα οι επαγγελματίε του χρηματοπιστωτικού κλάδου, αλλά να υπάρχει μια εξισορρόπηση των διαφόρων συμφερόντων. Και είναι ακριβώς αυτό το Εποπτικό Συμβούλιο το οποίο εποπτεύει τα κριτήρια επιλογής των μελών του ISB. Είναι σημαντικό λοιπόν να συνεχίσουμε να έχουμε μια παρουσία σε αυτό το εποπτικό συμβούλιο για να μπορέσουμε να επηρεάσουμε τα τεκτενόμενα. Και πάντα φυσικά μπορούμε να επιφέρουμε βελτιώσεις στη διακυβέρνηση αυτών των οργανισμών και αυτό είναι το αντικείμενο ενός σχεδίου που έχουμε ξεκινήσει. Αλλά Πάντα θα πρέπει να ξέρουμε ότι το ISB έχει κάνει μεγάλη πρόοδο, Έχουμε, έχει περάσει από ένα μικρό φορέα, ο οποίο ήταν, όπω ελέγχθη, σχεδόν απόλυτα αγγλοσαξονικό, σε ένα διεθνή φορέα, ο οποίο είναι πολύ πιο διαφανής και αυτό υπογραμμίστηκε από τα μέλη τη Επιτροπής σα, και προς την κατεύθυνση αυτή και μέσα στο πλαίσιο αυτό η Κομισιόν παρουσίασε την τρέχουσα πρόταση. Βλέπω τώρα τα τις σημειώσεις μου μιλήσαμε για τη διαδικασία έγκρισης των προτύπων. Φυσικά έχει κεφαλαιόδη χαρακτήρα αυτή η διαδικασία και θα πρέπει να την επανεξετάσουμε μετά από τα πορίσματα της αξιολόγησης που θα ξεκινήσουμε και μετά από το πέρας της αποστολής του κ. Μέιστατ. Νομίζω ότι έχω καλύψει όλα τα θέματα. Ευχαριστώ πολύ και την Επιτροπή για τα σχόλιά της. Ο κύριος Γκίκορτ ήθελε πάλι το λόγο. Λοιπόν, ε, πολύ ενδιαφέρον. Στείλτε τις καλύτερες ευχές μου στον κύριο Μάιστατ. Πάντα είχα καλή εντύπωση όταν ερχόταν εδώ και ανταλλάσσαμε απόψει και έπαιξε καλό ρόλο. Άλλαξε κάποιες ε, ελλείψεις στον φάτη διαφάνεια. Αν καταφέρει όπως άλλαξε το ERB να αλλάξει και το ISB. E θα τον πάω να τα πιούμε κιόλα. Θα τον κεράσω. Θα με ενδιέφερε να ξέρω αν μπορείτε να μας πείτε εδώ στην Επιτροπή ποια εντολή του δόθηκε. Και ίσως θα μπορούσαμε να συζητήσουμε επικοδομητικά το θέμα μαζί του. Όλα τα θέματα που του δημοκρατικού ελέγχου και, όσο, και την πλήρη διαφάνεια για προπολογισμό, επιρροή κλπ αν όλα αυτά εμπίπτουν στην εντολή του. Θα ήθελα να το ξέρω. Και κατά πόσο, ανεξάρτητα από το αν είναι Αγγλοσάξον ή όχι, αυτό δεν είναι πρόβλημα για μένα. Κατά πόσο τα ευρωπαϊκά πρότυπα συμπεριλαμβάνονται σε αυτούς τους φορείς. Και τα, οι αγγλοσαξονικοί οργανισμοί έχουν ε, τα ίδια δημοκρατικά πρότυπα όπω τα ευρωπαϊκή φορείς. Ε, δεν είναι πρόβλημα. Το ISB είναι λίγο γερμανικό, λίγο τσεχικό, λίγο αμερικανικό, λίγο βρετανικό όσον αυτά τα πρότυπα. Δεν είναι μια δομή όμως που δημιουργήθηκε από παραδοσιακές δημοκρατικές αξίες και ο τρόπος πρόσληψης των μελών των φορέων λήψεως απόφασης γίνεται με τρόπο που δεν αντιστοιχεί σε θεσμούς ε, που παράγουν δημόσια αγαθά. Καλό είναι για ιδιωτικού φορείς. Αλλά είναι προβληματική αυτή η μέθοδος για κάποιο φορέα που υποτίθεται ότι λογοδοτεί όσον αφορά την παραγωγή δημοσίων αγαθών. Θα ήθελα να γνωρίζω περισσότερο όσον αφορά την ε, εντολή που δόθηκε. Ευχαριστώ κύριε Γκίγκολτς. Ο Στόλογιαν, θέλετε να προβείτε σε κάποιο σχόλιο. Ναι, λέει κύριος Ευχαριστώ Πρόεδρε. Υποτίθεται ότι θα άκουγα πολύ ενδιαφέροντα σχόλια όσον αφορά την έκθεση. Το ήξερα, ήμουν βέβαιος. Διότι χρειάστηκα πολύ χρόνο να καταλάβω τι έπρεπε να κάνουμε όσον αφορά αυτή την ε, έκθεση. Το πρόβλημα είναι ότι έχουμε δουλειά να κάνουμε, κάτι να κάνουμε όσον αφορά αυτή την έκθεση. Και υπάρχουν διάφορα ζητήματα που έχουν τεθεί εδώ. Συμφωνώ απόλυτα με αυτά που υπόθηκαν. Όμως, ο χρόνος για να βρεθεί απάντηση στα ζητήματα δεν αρκεί ε, όσον αφορά το χρόνο που έχει διατεθεί για την έκθεση. Κύριε Κλίνς, μιλήσατε για το Συμβούλιο που εποπτεύει τα δημόσια συμφέροντα. εποπτεύει τη Διεθνή Ομοσπονδία ε, Λογιστών. και άλλους φορείς ε, που είναι υπεύθυνοι για τον έλεγχο του τομέα. Ρωτήσατε εάν θα πρέπει να χρηματοδοτούμε ακόμα αυτό τον οργανισμό. Πρέπει να συνεχίσουμε τη χρηματοδότηση του φορέα. 2,3 εκατομμύρια μόλις είναι για μία επταετία. Το μικρότερο ποσό. Και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι ε, ε ιδρυτικό μέλος της ομάδας ελέγχου και δύο από τα δέκα μέλη στο PIOB έχουμε και θα πρέπει να είμαστε σε αυτόν τον οργανισμό, να είμαστε μέσα παρόντες. Έχουμε ανοίξει την πόρτα του οργανισμού και να κρατήσουμε το πόδι μας να παραμείνει και η πόρτα ανοιχτή, να είμαστε μέσα. Η συγχρηματοδότηση είναι 22% του συνολικού προϋπολογισμού και είναι το ίδιο ποσοστό όπως και στο προηγούμενο πρόγραμμα. Το 2011 το ίδιο ποσοστό συγχρηματοδότησης είχαμε, 22% του προϋπολογισμού. Με αυτό τον οργανισμό είχαμε αναλάβει μία δέσμευση στην προηγούμενη έκθεση. Μάλλον αυτοί είχαν αναλάβει υποχρέωση να έχουν ευρύτερο φάσμα όσον αφορά τις πηγές χρηματοδότησης. Διότι είχαν μόνο δύο πηγές. Διεθνής Ομοσπονδία Λογιστών, η μία πηγή και η Ευρωπαϊκή Ένωση η άλλη πηγή. Και στο προηγούμενο πρόγραμμα, πώς να το πω, είχαμε αναθέσει καθήκον σε αυτόν τον οργανισμό να βρει και άλλες πηγές χρηματοδότησης. Τους ρώτησα αν το έκαναν αυτό και φαίνεται ότι το κατάφεραν αυτό. Αυτά για αυτή την ερώτηση. Σχετικά με αυτό που είπε ο κύριος Γκίγκολ, την πρότασή του, να διεξαχθεί εδώ μια ακρόαση στην Επιτροπή μας. Να συμμετάσχει που αυτοί οι τρεις οργανισμοί. Αυτοί που χρηματοδοτούμε από τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, πολύ καλή ιδέα. Μπορούμε να το οργανώσουμε. Θα το συζητήσω με την κυρία Μπόλς Να διοργανώσουμε μια ακρόαση. Με κοιτάει, πώς με κοιτάει, με κοιτάει. Ε, δεν νομίζω να μην έχουμε λεφτά για κάτι τέτοιο. Δεν φαντάζω. Από τα 58 εκατομμύρια που θα τα εξοικονομήσουμε. Οπότε θα είναι τεράστια ακρόαση. Αν πάρουμε αυτά τα λεφτά. Συνεχίζω και ο Στόλογιαν. Το τελευταίο. Έχουμε ένα νέο καθήκον. Νέο σύμβουλο για τον Επίτροπο Μπαρνιέ. Και νέο καθήκον που ανετέθη στον κύριο Μάιστατ. Μέχρι τέλος Νοεμβρίου να υποβάλει έκθεση, να εμφανιστεί στην Επιτροπή ΕΚΟΝ και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μας πει τι πρέπει να γίνει για να βελτιωθεί η διακυβέρνηση όλων αυτών των οργανισμών και νομίζω ότι το αίτημα του κυρίου Γκίγκολτ το υποστηρίζω έναντι αυτού του Συμβούλου. Νέο αίτημα. Το ταχύτερο δυνατό να του ζητήσουμε να γίνει μια ανταλλαγή απόψεων στην ΕΚΟΝ, να έρθει εδώ και να ανταλλάξουμε απόψεις. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Στόλογιαν. Και τώρα το χρονοδιάγραμμα της έκθεσης. Το σχέδιο θα παρουσιαστεί στις 11 Απριλίου εφέτος. Η προθεσμία για τις τροπολογίες είναι 30 Απριλίου. Η συζήτηση για τις τροπολογίες θα γίνει στις 28 Μαΐου και η ψηφοφορία στην Επιτροπή Οικονομικών Θεμάτων στις 24 Ιουνίου. Στην Ολομέλεια δεν γνωρίζουμε ακριβώς πότε και έτσι έχουμε φτάσει στο τέλος Τη συνεδρίαση. Έχω να σας κάνω μια σημαντική ανακοίνωση για αύριο μονάχα. Ο οικονομικό και νομισματικό διάλογο με τον πρόεδρο του Eurogroup, τον κύριο Ντέισελ Μπλουμ, θα λάβει χώρα στη, στην αίθουσα 3 σε 050. Όχι σε αυτή την αίθουσα. Θα ήθελα να σα ζητήσω να είσαστε εγκαίρος στι 9 γιατί ο πρόεδρος Ντέισελμπλομ θέλει να, πρέπει να φύγει στις 10.30 ε, και εμείς πρέπει να ψηφίσουμε. Μέχρι αύριο.